Ο κύριος Τζοβάνι Τόκη ε, εξελέγει ε, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λιγουρίας από 10 Ιουλίου 2015 η θέση του χειρεύει. Τον συγχαίρομαι. Οι αυστριακές αρμόδιες αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή της ε, κυρίας Καρολίνας Γκρας Βάντερ Χάιντς που αντικαθιστά τον κύριο Γιώργ Λάιχτφριντ ε, από 9 Ιουλίου. Οι Ιταλικές αρμόδιες αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Στέφανο Μαουλού ε, από 13 Ιουλίου 2015 αντικαθιστά τον κύριο Τζοβανιτότη, Οι ελληνικές αρχές ε, μου ε, με ενημέρωσαν για την αντικατάσταση από τον κύριο Νικόλα Οχούντη, διού Εμμανουήλ Γλέζου από 20 Ιουλίου 2015. Οι αρμόδιες σουηδικές αρχές με ενημέρωσαν για την εκλογή του κυρίου Γιασέγκο Σελίμοβιτς ε, με ισχύ από 30 Σεπτεμβρίου 2015. Αντικαθιστά την κυρία Μάριτ Πάουσεν. Οι Ολλανδικές αρχές με, ενημερώ, με ενημέρωσαν για την εκλογή ε, του κυρίου Άουκερ Ζήλστρα που αντικαθιστά τον κύριο Χάνς Γιάνσεν με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2015. Καλωσορίζω τους συναδέλφους ε, και βεβαίως ε, συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με το καταστατικό